Τώρα μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη έκθεση της κυρίας Σφίκα. Το ευεργέτημα παινίας σε διασυνοριακές διαφορές επί αστικών και εμπορικών υποθέσεων. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή η έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας όσον αφορά την δικαστική αρρωγή σε διασνοριακές διαφορές επιαστικών και εμπορικών υποθέσεων ουσιαστικά απορρέει από την εφαρμογή της οδηγίας του 2003 Τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη βελτίωση τη πρόσβαση στη δικαιοσύνη επί διασυνοριακών διαφορών. Μπορούμε να πούμε ότι η οδηγία αυτή ήταν γενικά επιτυχη. Δυστυχώ όμω δεν την έχουν εφαρμόσει όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι το δικαίωμα δικαστική αρρωγή πάντω ε, το έχουν εγγυηθεί τα περισσότερα κράτη-μέλη. Παρ' όλα αυτά, 12 μόνο τις 100 των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενήμεροι για την ύπαρξη δικαστικής αρρωγής σε διασυνοριακές διαφορές. Αν λοιπόν οι ίδιοι πολίτες ε, και ακόμα χειρότερο ε, όσοι ασκούν νομικά επαγγέλματα δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει δυνατότητα δικαστικής αρρωγής σε διασυνοριακές διαφορές, τότε καταλαβαίνετε ότι οι διατάξεις της οδηγίες παραμένουν απλώς θεωρητικές. Η ε, αυξανόμενη κινητικότητα και εναρμόνιση της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδηγήσουν σε όλο και μεγαλύτερο αριθμό διαστοριακών διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, ο αριθμός των πολιτών που κάνουν αίτηση για δικαστική αρρωγή είναι ακόμα πολύ χαμηλός, ακριβώς επειδή οι περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτες, όπως σας είπα, δεν γνωρίζουν ακόμα ότι μπορούν να έχουν ε, δικαστική αρρωγή σε μια άλλη χώρα πέρα από την δικιά τους. Επομένω, δεν κάνουν ποτέ την ανάλογη αίτηση. Στην έκθεσή μου λοιπόν επικεντρώθηκα σε κάποια μέτρα και σε κάποιες εκστρατείες που θα μπορούσαν να ευαισθητοποιήσουν περισσότερο τους πολίτες ως προς τη δυνατότητα αυτή, δηλαδή τη χορήγηση δικαστικής αρρωγής. Επίσης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και κάποια νέα τεχνολογικά μέσα προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες για τα δικαιώματά τους σε διαστοριακές διαφορές. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η διαδικτυακή πύλη e-justice προκειμένου να καταφέρουν οι πολίτες να κάνουν αίτηση δικαστικής αρρωγής. Επίσης θεωρώ ότι θα πρέπει να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε και κάποιες βάσεις δεδομένων δικηγόρων, νομικών νομομαθών, οι οποίοι θα έχουν τις απαραίτητες γλωσσικές ικανότητες και θα γνωρίζουν κάποια στοιχεία συγκριτικού δικαίου και πολλές φορές και το δίκαιο άλλων χωρών. Κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν οι άνθρωποι αυτοί να αναλάβουν την διαχείριση περιπτώσεων δικαστικής αρρωγής σε διασυνοριακές διαφορές. Καταλαβαίνετε ότι δοθεί το καθήκον αυτών σε ανθρώπους οι οποίοι δεν θα είναι απαραίτητα κατερτισμένοι, θα είναι κάτι το ιδιαίτερο αντιπαραγωγικό. Επίσης αναφέρομαι σε κάποια βήματα τα οποία θα πρέπει να ελοποιηθούν προκειμένου να διευκολύνουμε την όλη διαδικασία και την πρόσβαση σε δικαστική αρρωγή. Ενθαρρύνονται λοιπόν τα κράτη-μέλη να εντείνουν τη συνεργασία ανάμεσα σε μη κυβερνητικέ οργανώσει και αρμόδιε κρατικέ αρχέ. Επίση, κάποιε βέλτιστε πρακτικέ στον τομέα τη δικαστική αρρωγή θα πρέπει να προωθηθούν ακόμα περισσότερο. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τη δραστηριότητα όλων αυτών των αρμόδιων εθνικών αρκών, οι οποίε θα πρέπει να αποτελέσουν τμήμα ενό γενικότερου ευρωπαϊκού δικτύου δικαστική αρρωγή. Διανύουμε δύσκολε οικονομικέ περιόδου, επομένω είναι πάρα πολύ δύσκολο πάρα πολύ σημαντικό, με συγχωρείτε, τα κράτη-μέλη να είναι σε θέση να δίνουν εκ των προτέρων τις απαραίτητες πληροφορίες για τη δυνατότητα χορήγησης δικαστικής αρρωγής, ιδίως στην περίπτωση των διασυνοριακών διαφορών. Ιδίως όσον αφορά βέβαια τις αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Πρέπει να σας πω ότι με ανησυχούν επίσης όλες οι περικοπές που έχουν γίνει στον προπολογισμό όσον αφορά την χορήγηση δικαστικής αρρωγής. Καταλαβαίνετε ότι, κάτι τέτοι, ότι τέτοιες δημοσιονομικές περικοπές ουσιαστικά δεν θα επιτρέψουν σε πάρα πολλούς πολίτες να έχουν πρόσβαση σε δικαστική αρρωγή και κατά αυτόν τον τρόπο θα οδηγήσουν και στην, στην, στο να καταλήξουν οι πολίτες σε μια πιο δυσχερή κατάσταση τελικά. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή. Διαδικασία Catch the Eye. Η Μαρή Τερέση Σάντσες έχει το λόγο. Α, συγγνώμη, εγώ νομίζω ότι ήμασταν ήδη στο επόμενο θέμα. Τότε θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο. Α, ο κύριος Πλάτς, ζητήσατε το λόγο. Έχετε το λόγο. Θα είμαι ο μόνος ο μιλητής για αυτό το θέμα από ό,τι φαίνεται, αλλά επιμένω διότι θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα και ευχαριστώ τον συνάδελφο που το πραγματεύτηκε στην έκθεσή του, διότι ε, στο, θα μπορούσαμε να αυξήσουμε, λέει ο μιλητή, την ανταγωνιστικότητα στο διασυνοριακό εμπόριο. Μπορούμε να τονίσουμε επίση τη σημασία με, ε, ε, της συνεργασίας με τα τεχνικά επιμελητήρια. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντικό να γνωρίζουν ότι δικαιούνται ευεργέτημα παινίας στις διασυνοριακές περιπτώσεις και ότι δικαιούνται νομική αρρωγή για την εκδίκαση μιας υπόθεσης που τους αφορά. Υποστηρίζω επίσης την ιδέα της ε, βάσης δεδομένων ε, δικηγόρων με τις κατάλληλες γλωσσικές ε, δεξιότητες. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να τονίσω προς όλους τους ομιλητές ότι πρέπει να μιλάμε για το σημείο της ημερήσιας διάταξης που εξετάζουμε και αν επιθυμείτε το λόγο θα πρέπει εγκαίρως να το δηλώνετε. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε ρωτήσουμε λοιπόν, έτσι θα διευκολυνθεί η διεξαγωγή της συζήτησης. Σας δώσουμε τώρα το λόγο στον Επίτροπο. Thank you, Mr. President, honorable members. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική του αυτή έκθεση και για το ότι ανέκαθεν υποστήριζε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταρρύψει οποιαδήποτε εμπόδια υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην παροχή δικαστικής αρρωγής σε διασνοριακές διαφορές για τους Ευρωπαίους πολίτες. Το μέσο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα επιτρέψει στους Ευρωπαίους πολίτες να καταφέρουν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους προσφυγής σε δικαστικά συστήματα άλλων κρατών μελών. Έχουμε όντω την οδηγία του 2003-8 για την βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη επί διασυνοριακών διαφορών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε ήδη μια έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας αυτής και αναφέρεται σε όλες αυτές τις χώρες οι οποίες έχουν μεταφέρει την οδηγία αυτή. Δεν έχουμε εντοπίσει σημαντικά προβλήματα στην ε, εφαρμογή της οδηγίας αυτής, μόλον ότι ακόμα υπάρχουν διαφορές, διαφορε, διαφορές ερμηνείας από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Το γεγονός ότι είχαμε μόνο μία περίπτωση προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όσον αφορά δικαστική αρρωγή σε διασυνοριακές διαφορές καταδεικνύει ότι η εφαρμογή της οδηγίας από νομικής πλευράς είναι ικανοποιητική. Ωστόσο, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η γνώση των ίδιων των πολιτών αλλά και των δικηγόρων για τα ευεργετήματα τη οδηγία αυτή δεν είναι επαρκή. Επομένω, θα πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλει ήδη προσπάθειε ω προ αυτό. Προσπαθούμε να επικαιροποιήσουμε την διαδικτυακή πύλη e-Justice προκειμένου να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση των πολιτών και πιο τυποποιημένη παροχή πληροφόρηση. Επίσης, η αντίστοιχη ιστοσελίδα για το διαδικτυακή πύλη e-Justice θα βελτιωθεί προκειμένου να δοθούν πιο επικαιροποιημένε και βελτιωμένε πληροφορίε προ πολίτε. Κατά αυτόν τον τρόπο θα ενημερώνονται οι πολίτε με πολύ καλύτερο τρόπο και για άλλε διαδικασίε όπω η διαδικασία, ευρωπαϊκή διαδικασία αποζημίωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε την χορήγηση δικαστικής αρρωγή σε διασυνοριακές διαφορές επιαστικών και εμπορικών υποθέσεων. Ήδη έχει συνταχθεί ένα εγχειρίδιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο έχει δοθεί σε νομικούς και νομαθεί σε διάφορες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωση. Είχαμε μιλήσει και στο παρελθόν για την οδηγία αυτή και είχαμε πει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εφαρμόζεται σε όλε τι χώρε. Θα πρέπει όμω να καταφέρουμε να, να βοηθήσουμε του δικηγόρου να συνειδητοποιήσουν ποια είναι τα ωφέλη τη οδηγία αυτή και να ενημερώσουμε καταλήλω και του πολίτε. Είναι πολύ σημαντικό ένα πιλωτικό πρόγραμμα για την κατάρτιση των δικηγόρων να υλοποιηθεί. Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθούν και πλατφόρμες κατάρτισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τους νομομαθείς. Στο επόμενο, στην επόμενη χρηματοδοτική περίοδο προβλέπονται τα απαραίτητα κονδύλια για να βοηθήσουμε στους τομείς αυτούς τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά τώρα το ρόλο που μπορούν να δραματίσουν τα κράτη-μέλη, όπως είπατε, όπως είπατε και εσείς στην έκθεσή σας, είναι πολύ σημαντικό να ενημερώσουν τους πολίτες τους για τα δικαιώματά τους στα πλαίσια της οδηγίας αυτής και για τα όσα προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία. Η πρότασή σας, η εκθέσή σας μάλλον προβλέπει πολλές προτάσεις τροποποίησης της οδηγίας, καθώς επίσης και κάποιων στοιχείων που θα μπορούσαν να προστεθούν στην οδηγία. Θα λάβουμε λοιπόν υπόψη τις προτάσεις αυτές στην εργασία που θα επιτελέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τομέα αυτό στο μέλλον. Είναι πολύ σημαντικό να επικεντρωθούμε περισσότερο στην καλύτερη ενημέρωση των πολιτών για τα δικαιώματά του και στην καλύτερη παρακολούθηση τη εφαρμογή οδηγία αυτή από τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη όταν ζητήσαμε την άποψή του για την οδηγία αυτή μα είπαν ότι δεν θεωρούν ότι θα πρέπει να γίνει κάποια τροποποίηση τη οδηγία. Επομένως, οποιαδήποτε δράση αναλυφθεί σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο θα πρέπει να έχει ως στόχο την καλύτερη προώθηση της οδηγίας και την καλύτερη παροχή επικαιροποιημένων πληροφοριών για τις δυνατότητες δικαστικής αρρωγής προβλέπονται σε κάθε κράτος μέλος. Θεωρούμε ότι κατά αυτόν τον τρόπο όλο και περισσότερες πολίτες θα έχουν πρόσβαση στο δικαίωμα αυτό, όπως περιγράφεται άλλωστε στο άρθρο 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης zu diesem Tagesordnungspunkt. Όσον αφορά την ψηφοφορία για αυτό το σημείο τη σημερινή διάταξης θα λάβει χώρα αύριο στις 11 και 30. Και τώρα περνάμε στην έκθεση του Αντιπροέδρου Πλάσακ όσον αφορά την περιφερειακή πολιτική ως μέρος ευρύτερων κρατικών